Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει με την ολοκλήρωση των συζητήσεων το απόγευμα. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση για τον Μπαχρέιν και συγκεκριμένα τις περιπτώσεις Ναμπίλ Ρατζάμπ, Αμπτουλ Χατί Αλ Καουάια και Ιμπραήμ Σαρίφ. Συντάκτες με τον κύριο Κέλλαν πρώτο για ένα λεπτό. Τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ισορροπημένη και επικοδομητική προσέγγιση που θα συνδυάζει και κριτικό όμα και ενθάρρυνση. Ε, υπάρχουν λόγια να ανησυχούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο στο στον Μπαχρέιν και για την καταστολή τα τελευταία χρόνια των διαδηλώσεων. Και σήμερα σαφώς ζητούμε να απελευθερωθούν διάφοροι φυλακισμένοι κρατούμενοι συνειδήσεις, ο Ραμπέλ Ρατζάμπ, Αμπτούλ Χάντι, Κουάλτσα και ταυτόχρονα νομίζω ότι υπάρχουν και ενθαρρυντικά σημάδια ότι η κυβέρνηση του Μπαχρέιν έχει αναλάβει την υποχρέωση να κάνει μεταρρυθμίσεις. Με, σύμφωνα με την, εξάρτητη, την έκθεση της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ερεύνης του Μπαχρέιν και θα γίνονται και προσπάθειες ε, αναδιαμόρφωσης του ποινικού κώδικα, ούτως ώστε τελικά η δικαιοσύνη να γίνει ανεξάρτητη. Και υπάρχει και ξεκίνησαν διάλογοι με τον ε, πρίγκιπα, με τον διάδοχο πρίγκιπα. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, θα εκφράζουμε κριτική, αλλά πρέπει να ενθαρρύνουμε τις αρχές του Μπαχρέιν να κάνουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε Κίλαμ. Βαν Όρντεν, συνάδελφος Βαν Όρντεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλωσορίζω το τα σχόλια του κυρίου Κίλαμ και την έκθεση γενικά που είναι πολύ ισορροπημένη. Βέβαια, Πρέπει να στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να βοηθούμε τους άλλους στο μονοπάτι των μεταρρυθμίσεων. Πρέπει να αναγνωρίζουμε και την πραγματικότητα που ισχύει σε κάθε περίσταση. Η παρουσία κρεφνών στοιχείων, παρέμβαση από άλλες χώρες που θέλουν να αποστεθεροποιήσουν ένα καθεστώς και βέβαια την ανάγκη για νόμο και τάξη. Αλλά αυτό από μόνο του δεν αποτελεί εξουσία για αυθαίρετη φυλάκιση. Το Μπαχρέν είναι μια χώρα που μακρόν ήταν φίλος και σύμμαχος της δύση και ιδιαίτερα της χώρας μου. Μετά από πρωτοβουλία του Βασιλέως, ο διάδοχος του Μπαχρέιν ε, έδειξε μεγάλες ηγετικές ικανότητες ε, για επιβολή μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν τη δημοκρατία και θα βοηθήσουν την επίτευξη σταθερότητα. Όλοι, οι πρόθυμοι, με καλή, καλή βούληση πολιτική στον Μπαχρέιν εξάρτητα κόμματο, θα πρέπει επικοδομητικά να συμμετάσχουν στον εθνικό πολιτικό διάλογο και οι αρχές του Μπαχρέιν από την πλευρά τους θα πρέπει να δείξουν αυτοσυγκράτηση και γενεοδορία όσον αφορά αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Κύριε Βανόρντε, δεχόσαστε από τη συνάδελφο Σάλκε μια ερώτηση. Δεχόσαστε. Κυρία Σάλκε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. δε κύριε Σάκε. Με τα χαρά άκουσα κύριε Βαν Όρντερ ότι ανησυχείτε και εσείς με παρεμβάσεις από εξωτερικούς φορείς όπως είναι το Ιράν και η Σαουδική Αραβία. Η ομάδα μας ε, πρότεινε να αναφερθούν αυτές οι ανησυχίες στο ψήφισμα, αλλά η δική σας ομάδα, όπως και το ΕΛΚ, δεν θέλα να γίνει αυτή η μνήμα. Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε την ευρύτερη εικόνα στο, στη Μέση Ανατολή για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα στον Παχρέν και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα, διότι έχουμε χειρότερε κρίσει να αντιμετωπίσουμε. Ήθελα να ρωτήσω, συμφωνείτε ότι πρόκειται περί προβλήματος που πρέπει να μα απασχολεί. Ο κ. Βανόρντεν. Όπως, ο καλός, όπως ξέρετε η, καλή συνάδελφος δεν αναφερόμουν στην Σαουδική Αραβία με αυτά που είπα. Η Σαουδική Αραβία είναι φίλη και σύμμαχος του καθεστώτος. Εγώ αναφερόμουν σε παρεμβάσεις από χώρες από την άλλη πλευρά του κόλπου και κυρίως από το Ιράν. Ευχαριστώ κύριε Βανόρντεν. Για δύο λεπτά, κυρία Δεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τα ψηφίσματα της πέμπτης απόγευμα δεν θα πρέπει να είναι αντιπαραγωγικά. Ιδιαίτερα για μια χώρα με τόσο ευαίσθητη κατάσταση όπως είναι το Παχρέιν με αντιπαράθεση συνητών, σουητών και, και σουνητών. Ε, φυσικά θα πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα οι εκτιβιστές. Ε, χαιρετίζουμε τις προσπάθειες επανασυμφιλίωσης του διαδόχου του θρόνου. Έχουμε την τρίτη επέτειο της εξέγερσης στον Παχρέν και εδώ και τρία χρόνια η καταστολή δυστυχώς έχει μείνει αμύωτη. Η... Πολλοί διεθνεί εταίροι και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησαν περισσότερη δημοκρατία και άνοιγμα τη χώρα αυτή. Αλλά 15 Ιανουαρίου ο διάδοχο ε, έκανε ένα βήμα πρόοδου, άνοιξε το, τον, διάλογο, τον Εθνικό Διάλογο Επανασυμφιλίωσης, όρισε διαμεσολαβητή στο Υπουργείο Εσωτερικών, μια ειδική επιτροπή ερευνών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και επίσης ε, μια επιτροπή που θα ενημερώνει και θα καταγγέλει περιπτώσεις ε, ε, κακοποίησης των κρατουμένων. Όλα αυτά είναι θετικά βήματα. Αυτά όμως τα σχέδια θα μπορούσαν να είναι ένα απλό παραπέτασμα καπνού για να κατα κατευναστεί η παγκόσμια κοινή γνώμη. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση στο Μπαχρέιν, στηρίζοντα του μεταρρυθμιστέ που θέλουν με ειρηνικό τρόπο να μεταμορφώσουν και να μεταρρυθμίσουν τη χώρα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κυρία Τεκεζέχ. Για δύο λεπτά η κυρία Βεργιά. Το Μπαχρέιν μαστίζεται ακόμη από μια βαρύτατη καταστολή Τρία χρόνια τώρα δεν ε, επιτρέπεται η έκφραση καμία ε, αντιφρονούσα γνώμη στο ιστορικό στο εξωτερικό. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Γνωρίζουμε τι είδου ε, διακυβεύματα υπάρχουν, τι υπάρχει, τι προοδεύει, τι οπισθοδρομεί, τι, τι παραμένει στάσιμο. Έχουμε παρακολουθήσει την χρήση διαφόρων μέσων συμπεριλαμβανομένου και αυτού ε, της απόπειρας να μας κάνουν να πιστέψουν ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ σύντων. Παραμένει λοιπόν ε, σκοτεινή αυτή η άνοιξη της, ε, του Μπαχρέν, η οποία δυστυχώς επισκιάστηκε χάρη στις, ε, στην υποστήριξη προς το καθεστώς των αρα, των Σαούδων εξαδέλφων. Δεν μπορεί λοιπόν να προχωρήσει η χώρα αυτή παρά μόνο μένει στα χέρια αυτού του καθεστώτος το οποίο με κάποια ανταλλάγματα εξασφαλίζει την υποστήριξη των δυτικών δεν μπορούν οι αντιφρονούντες να εκφράσουν τις θέσεις τους. Είναι 3.000 οι πολιτικοί κρατούμενοι σε μια μικρή χώρα με 600.000 κατοίκους. Όλοι γνωρίζουν ότι δεν κυβερνά ο πρίγκιπς στον Μπαχρέιν, αλλά ο Πρωθυπουργό εδώ και 50 χρόνια, ο θείο του. Η ελευθερία της έκφρασης παραβιάζεται συστηματικά για τους εθνικούς αλλά και για τους εγχώρους αλλά τους ξένους δημοσιογράφους. Η χώρα αυτή έχει κηρύξει πόλεμο στο ίντερνετ δεν επιτρέπει ούτε μία αμφισβήτηση εξουσίας. Θέλω να αναφερθώ στον Αμπίλ Χαρατζάμπ, πρόεδρο της ε, Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα στο Μπαχρέιν και αντιπρόεδρο της Διεθνούς Οργανώσης και τον Αμπτουλ Χαντί Αλκαουάια, που ε, βασανίστηκαν ε, σκληρά και έμειναν στη φυλακή, έχουν καταδικαστεί ισόβια δεν υπάρχει καμία ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον οργανισμό για τη συνεργασία στον Περσικό. Αυτό τα λέει όλα νομίζω και το γεγονός ότι το Μπαχρέ είναι από τους κύριους αγοραστές όπλων, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες παρουσιάζει μεγάλη έμφαση, δεν αποτελεί καλό ιονό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάκε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι οι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα αρχέ των Μπαχρέιν δεν θα επισκιαστούν από διαφημιστικέ εκστατείε ή υποχορηγίε ε, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο CNN. Όποιο δει εκ του σύνεγγυ τι γίνεται στο Μπαχρέιν καταλαβαίνει ότι είναι μια ντροπή που η βασιλική οικογένεια και η κυβέρνηση δεν κατάφεραν επαρκώ να αντιμετωπίσουν ανησυχίε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διαμαρτυρίες και τις ανησυχίες του λαού. Να τονίσω ότι δεν χρειάζονται επανέμβαση από κα... ούτε από τη Σαουδική Αραβία ούτε από το Ιράν όσον αφορά τα εσωτερικά του ζητήματα. Ανταυτού η έκθεση καθώς και διάφορες συστάσεις που γίνονται θα πρέπει να εφαρμοστούν τελεία και παύλα. Εντοπίσαμε και κάποιες άλλες κατεπίγους μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να λάβουν χώρα οι εξαφανίσει είναι κάτι που καταγγέλουμε και η χρήση στατοδικείων και ειδικών δικαστηρίων να ε, δικάζουν αυτούς που θεωρούνται ύποπτοι για εθνικά εγκλήματα. Δεν θα πρέπει οι γιατροί να εμποδίζονται και θα πρέπει να κάνουν την ε, δουλειά τους, κυρίω όσον αφορά του νέου κρατουμένου, του ανήλικου, θα πρέπει τον να τους μετωπίσει σύμφωνα με του κανόνε του ΙΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, διότι έχει υπογράψει αυτό το ε, σύμβαση τον Μπαχρέιν. Και ζητάμε στο ψήφισμα για να πάγουμε όσον αφορά τη θανατική ποινή και ελπίζουμε τελικά η θανατική ποινή να καταργηθεί. μαχητέ, όπω ο Αμπτουχαντή Αλχαουάτζα και η κόρη του η Ζαϊνέπ δεν έχουν απελευθεί που είναι μαχητέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε Ρατζάμπ, ούτε Ιμπραήμ Σαρίφ. Για μία ακόμη φορά ζητούμε για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των ε, μαχητών για, την, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των πασπιστών των ανθρώπινων δικαιώματα. Και ελπίζω ότι η απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου να δημιουργήσει ένα δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι ένας καταλήτης που θα υπενθυμίζει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να σωτεύονται και στον Μπαχρέιν αλλά και σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Διότι το θλιβερό ποιο είναι. Βλέποντα τη Μέση Ανατολή, θα ήλπιζε κανεί ότι τα προβλήματα του Μπαχρέιν είναι που μπορούν να επιληθούν, θα αντιμετωπιστούν άπαξ διαπαντό. Ούτω ώστε οι φιλοδοξίε του για την θέση του στο παγκόσμιο προσκήνιο να μην είναι οικονομική φύσεω ή θετική φύσεω μόνο, αλλά θα πρέπει να δοθούν δικαιώματα και δυνατότητε και στο λαό του Μπαχρέιν. Έτσι και εγώ, σαν Ευρωβουλευτή, να μπορώ μπορώ να επισκεφτώ τη χώρα χωρίς να μου ε, αρνούνται την θεώρηση ευατηρίου. Ευχαριστώ κύριε Σάκε. Κύριο Σλούτερ, τελευταίο συντάκτη, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να ενθαρρύνουμε το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία να μην επεμβαίνουν στα εσωτερικά του Βαχρέιν. Αλλά δεν θα πρέπει το ίδιο να κάνουμε κι εμείς. Γιατί και εμείς κάνουμε εξαγωγές όπλων ή εθελοτυφλούμε δεχόμαστε προς τα... Ε, εθελοτυφλούμε δεχόμαστε την α ή β συμπεριφορά. Δεν είναι και αυτό ένα είδος επέμβασης ε, στα εσωτερικά του Μπαχρέιν. Δεν νομίζω ότι το διαδίκτυο απειλεί την ασφάλεια στον Μπαχρέιν. Και οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θέλουν απλώς να ασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης, εκ, ελεύθερης έκφρασης, ούτε και αυτοί απειλούν την ασφάλεια του Μπαχρέιν. Περισσότερο η ένοπλοι φρουροί του ε, βασιλικού οίκου απειλούν την ε, ασφάλεια του Μπαχρέιν. Αυτοί εμποδίζουν την ανοιχτή συζήτηση, το διάλογο και παρεμποδίζουν τη δημοκρατία. Η δημοκρατία απειλείται από την ε, διατήρηση της θανατικής ποινής και από την διατήρηση των ειδικών δικαστηρίων ή των στρατοδικείων. Αυτές είναι οι απειλές για το μέλλον του Μπαχρέιν. Θα πρέπει να γυρίσει σελίδα η χώρα αυτή και να εφαρμόσει ένα νέο σύστημα όχι να φυλακίζει τους επικριτές του καθεστώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σλίτλερ. Τώρα έχουμε τους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων. Ένα λεπτό κυρία Κόρχολα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Αντιμετωπίσαμε την κατάσταση επανειλημμένα στον Παχρέν στο Κοινοβούλιο τους τελευταίους μήνες και δεν το κάνουμε αυτό εις μάτιν. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια προβλήματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης το Μπαχρέιν είναι σε 25η θέση ε, όσον αφορά την ελευθερωτυπία. Και υπάρχουν μόνο 66 θέσει. Προτελευταία θέση. 44 δημοσιογράφοι και 22 μέλη των άλλων μέσων ενημέρωσης έχουν εμποδιστεί από το να ασκήσουν το επάγγελμά του. και η χρήση των κοινωνικών μέσων έχει εμποδιστεί. Μπορεί να φυλακιστεί Κανεί για πέντε χρόνια ή να πληρώσει πρόστιμο 10.000 ευρώ αν παραβεί την νομοθεσία. Μετά την έκθεση τη επιτροπή, ερευνητική επιτροπή του Μπαχρέιν, οι αρχέ υποσχέθηκαν να δράσουν, αλλά απομένουν πολλά που πρέπει να κάνουν οι αρχέ για να αποκατασταθεί η ομαλότητα σε αυτού του τομεί. Τα δικαστήρια δεν σέβονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζω ότι η δημιουργία αυτού του νέου δικαστηρίου θα έχει ε, ενεργη... Ε, θετικό αποτέλεσμα τελικά. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κόρχολα. Κύριο Στρέπφο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ζωφερή στο Μπαχρέιν. Οι αρχές επιβάλλουν απαράδεκτα μέτρα για να καταστήλουν διαδηλώσεις, δημαρτυρίες, για να καταστήλουν την έκφραση τις γνώμες. πολύ από τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετώπισαν μακροχρόνιες ε, ποινές κράτησης. Η χαλιναγώγηση λοιπόν της ελευθερίας ε, της έκφρασης ε, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης πρέπει να απαγορεύεται και πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη έκφραση για όλους τους κατοίκους του Μπαχρέιν, όπως βέβαια και σε όλο τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε φωνή στο λαό. Ο διαλόγος, ο εθνικός διάλογος πρέπει να πάρει προτεραιότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρέμβει σε μια κατάσταση απαράδεκτη που επικρατεί στο Μπαχρέιν. Η κατάσταση εκεί είναι απαράδεκτη, ιδιαίτερα στις φυλακές και πρέπει το χείτερο δυνατόν να αποφυλακιστούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρέπο. Κύριος Πόσλτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εκπροσωπώ την κυρία Νίπλερ ως πρόεδρο της αντιπροσωπείας για τα κράτη του Περσικού. Μας ανησυχεί η κατάσταση στο Παχρέν και βεβαίως και αγωνιζόμαστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως και απαιτούμε στις τρεις αυτές συγκεκριμένε περιπτώσεις πολιτικών κρατημένων να αναλάβουν το χειρότερο δυνατό δράση οι αρχές. Δεν μπορούμε όμως να συζητούμε με τόσο με νομερείς τοποθετήσεις όπως ακούσαμε από ορισμένου εδώ. Ε, πρώτα απ' όλα, εγώ έχω πρώτες αναμνήσεις εδώ και 30 χρόνια από την ανάληψη εξουσίας ε, του τωρινού ηγεμόνα στο Μπαχρέιν. Τακτονικές ε, πλάκες κινήθηκαν μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, τα προβλήματα με την περιοχή του ε, Ιράν, την προσπάθεια για επικοδομητικό ρόλο στην χώρα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή στην οποία και ο ηγεμόν αλλά και ο πρίγκιπας διάδοχος προσπαθούν να υποστηρίξουν. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για πιο αντικειμενική προσέγγιση στην περίπτωση του Μπαχρέιν και βέβαια προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Έτιγκερ. Ευχαριστώ. Η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέν δημιουργεί ε, τεράστιε ανησυχίε στη διεθνή ε, κοινή γνώμη. Φαίνεται ότι οι ε, αρχέ αγνοούν επιδεικτικά τις στοιχειώδεις ε, πολιτικές ελευθερίες όπως το δικαίωμα του συνέχιση και την ελευθερία έκφρασης θύματα άδικων συλλήψεων πέφτουν και δημόσια, δημόσια πρόσωπα όπως ο Ναμπίν Ρατζάβ που βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια στη φυλακή, είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Μπαχρέιν ή ο Αμπτουρχαντή Αλκαβάζα που είναι ακτιβιστής και που καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη για την ειρηνική του δραστηριότητα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ο Μπεραχήμ Σαρίφ γνωστός αντιφρονών του Μπαχρέιν που βρίσκεται στη φυλακή για συμμετοχή σε φιλελληνικές διαδηλώσεις το 2011. Αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και δεκάδε άλλοι που είναι θύματα αδιαφανών διαδικασιών, πλαστών αποδείξεων, εξευτελισμού βασανιστήριων και απάνθρωπη συμπεριφορά. Οφείλουμε να στυλιτεύσουμε την πολιτική αυτή και ζητούμε να εφαρμοστούν οι διατάξει τη έκθεση τη Ανεξάρτητη ε, Ερευνητική Επιτροπή του Μπαχρέιν του 2011 που καταδεικνύουν παράβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απάνθρωπη συμπεριφορά κατά των κρατουμένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία ο Έντινμπεργκ. Δεν θα κάνουμε διαδικασία καρουσία, δεν έχει στήσει κανεί το λόγο και έτσι δίνω το λόγο απευθεία στον Επίτροπο Φιούλα, Εκ μέρου τη Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, θέλω καταρχά να υπογραμμίσω ότι είπατε εκπρόσωπο και αντιπρόεδρος παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ στην κατάσταση στο Μπαχρέιν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει με τις αρχές επιτόπου επαφές σε κάθε επίπεδο και στο υψηλότερο, αλλά και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από την αναζωογόνηση των ταραχών το Φεβρουάριο πέρσι. Η Είπατε εκπρόσωπος καλωσορίζει τις ε, ειδήσει ότι ο διάδοχος κατά κατά του βασιλέος Αχμάτ έχει αναλάβει μια διαδικασία διαλόγου με, τον, με διάφορους εκπροσώπους κοινών πολιτών και με τον Σέικ Αλι Αλμάια από την πρώτη φορά που εμφανίστηκαν οι ταραχές το 2011. Σε αυτή τη, κρίση τη κρίσιμη λοιπόν συγκυρία πιστεύουμε ότι οι διαβουλεύσεις μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για μια μακροπρόθεσμη εθνική συμφιλίωση και βιώσιμη μεταρρύθμιση στο Μπαχρέιν. Απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις πλευρές να απόσχουν από τη βία και να συνεργαστούν μεταξύ τους για μια συμφιλίωση άνευ όρων. Όπως όμως είπαμε και επιμόνως τονίζουμε όλα αυτά τα χρόνια μια μακροχρόνια διαδικασία συμφιλίωσης χρειάζεται επίδειξη με τριοπάθειες και συγκεκριμένα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη από κάθε πλευρά, συμπεριλαμβανομένης και της αποφυλακής εκείνων που συνελήφθησαν στο πλαίσιο συμμετοχής τους ή λόγω συμμετοχής τους σε ειρηνικές ε, ε, διαδηλώσεις. Πρέπει να επανέλθει λοιπόν η ειρήνη στο Παχρέινο. Ο Σταύρος Λαπρινίδης, υπότιτλος εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, επισκέφθη τον Παχρέν τον Ιούνιο του 2013 και είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ορισμένους ε, πολιτικούς κρατουμένους, κρατουμένους για λόγους πολιτικών δραστηριοτήτων και μπορούμε να παρακολουθήσουμε ακόμη περισσότερο και πιο στενά τις ε, εξέλιξη στην υπόθεση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλωσορίζει τα σημαντικά βήματα που έχουν αναλάβει οι αρχές του Παχρέν για την υλοποίηση των συστάσεων της Ανεξάρτητης Επιτροπής Ερευνών του Μπαχρέιν, BICI, βελτιώνοντας έτσι την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αλλά πολλά ακόμα μένουν να γίνουν και πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε το Μπαχρέιν να εφαρμόζει σωστά και ταχύτατα την ε, τη συστάση του BICI, της Επιτροπής αυτής, Ανεξάρτητης Επιτροπής, αλλά και της ε, περιοδικής εκθέσεως των ΗΠΑ και θα συνεχίσουμε τις επαφές με τις αρχές ως προς την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ατιμορρησία και το ζήτημα της λογοδοσίας δεδομένου ότι και το Υπουργείο των Ιστορικών και ο Ομπουτσμαν και οι ανεξάρτητες αρχές και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι εκπρόσωποι των πολιτικών κρατουμένων και οι εκπρόσωποι των ε, οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να διαδραματίσουν σαφή και πρωταγωνιστικό ρόλο στην, στο πράσινο του για την ε, πρόοδο στην υπόθεση αυτή. Τα θεσμικά αυτά όργανα, οι θεσμοί αυτοί θα πρέπει να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για την ανάκτηση και της εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο κύριος Χουάν Μπεντέ, ειδικό απεσταλμένος στο Ηνωμένων Αθηνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασανιστήρια και τις απάνθρωπες, ε, την ανθρώπινη μεταχείριση στις συνθήκες κράτησης, ε, έχει όλη μας την υποστήριξη στην προσπάθειά του για καταγραφή των προόδων και θα ήθελα ιδιαίτερα να χαιρετήσω κλείνοντα τη συμβολή της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Αραβική Χερόνησο και να εκφράσω τις, την εκτίμησή μου για τις προσπάθειες που, που καταβάλει αυτή η αντιπροσωπεία, ιδιαίτερα σε σχέση με το Παχρέν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Φιούλε. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση κατατίθενται έξι ψηφίσματα. Τελειώνουμε εδώ τη συζήτηση και γίνεται ψηφοφορία αμέσως. Τώρα ξεκινούμε με τις ψηφοφορίες λοιπόν. Με πρώτο το θέμα της κατάστασης στην Ταϊλάνδη. Μία ψηφοφορία για ένα ψήφισμα κοινό πέντε ομάδων χωρίς τροπολογίες. Τελική ψηφοφορία λοιπόν υπέρ. Κατά.